και συνεργασία μέσα στα πλαίσια του ορίζοντα 2020. Πώς δηλαδή να δημιουργήσουμε πάνελς από κάτω προς τα πάνω και να υπάρξει και συνεργασία σε επιστημονικό επίπεδο. Ένα άλλο θέμα είναι το εύρος εφαρμογής από και για την κοινωνία. Σχετικά με τα θέματα Αυτά. Χρειάστηκε το Κοινοβούλιο να προχωρήσει περισσότερο. Ετοιμάσαμε λοιπόν κάποια έγγραφα για να διευκρινίσουμε και να αναπτύξουμε παρετέρω την θέση μας. Τη θέση που αναπτύξαμε και εδώ στην Επιτροπή αυτή τον Νοέμβριο που μας πέρασε. Δώσαμε δηλαδή επεξηγήσεις για την θέση μας αυτή. Τέλος, επιτρέψτε μου να σας πω ότι ακόμα Στου τριμερεί διαλόγους δεν έχουμε αγγίξει το θέμα του προπολογισμού. Εμεί, οι εισηγητέ και σκιώδες εισηγητέ, είμαστε απογοητευμένοι, όπω και οι περισσότεροι συνάδελφοι, όσον αφορά το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο και τη στάση που κράτησε το Συμβούλιο. Στόχος μας είναι ένα πιο ισχυρό πρόγραμμα ορίζοντας 2020 που να προσφέρει πραγματική ανάπτυξη και απασχόληση. Προς το παρόν δεν έχουμε βέβαια το τελικό ποσό, το τελικό κονδύλι για τον ορίζοντα 2020. Έχουμε για το ΣΑΤΛ 1α. Δεν έχουμε όμως την κατανομή ανάμεσα στο πρόγραμμα αυτό, το Εράσμους και διάφορα άλλα. Βέβαια, Μιλάμε για κάτι ανάμεσα στα 71 και 74 δισεκατομμύρια, ανάλογα με τον υπολογισμό που κάνει κανείς. Αυτή είναι η εκτίμηση. Ελπίζουμε να έχουμε σαν αποτέλεσμα ένα πιο φιλόδοξο ποσό, ένα πιο φιλόδοξο κονδύλι τώρα που έχουν αρχίσει οι διαπραγματεύσεις. Και ελπίζουμε να έχουμε έναν προϋπολογισμό, ο οποίος να τα αποκρίνεται καλύτερα στις φιλοδοξίες μας. Το πρόγραμμα αυτό είναι μία φιλοδοξία μας και ελπίζουμε να πρικοδοτηθεί κατάλληλα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Μαρία. Τώρα ο Ιβο Μπελέτ έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Πρόεδρε, θέμα όσο γίνεται πιο σύντομος. Έχουμε φτάσει σε μια ευρεία συμφωνία. Και έχουμε και ευρεία στήριξη της συμβαστικής αυτής θέσης με το Συμβούλιο μετά από πρώτη ανάγνωση και σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε για τον τόσο καλό τρόπο με τον οποίο προεδρεύσατε τη συνάντηση αυτή. Επίσης δεν πρέπει να ξεχάσω να πω ότι η πρόταση κανονισμού άλλαξε και έγινε πρόταση για οδηγία. Κάτι το οποίο είναι κεφαλαιόδου σημασία. Ένα από τα κύρια στοιχεία που στηρίξαμε είναι η ανεξαρτησία της αρμόδιας αρχής, που είναι ζωτική σημασία για το Κοινοβούλιο. Να υπάρχει δηλαδή διάκριση ανάμεσα στο διοικητικό σώμα στα κρατημέλη, το οποίο είναι αρμόδιο για την ασφάλεια των δράσεων και από την άλλη μεριά να έχουμε το διοικητικό εθνικό σώμα, το οποίο είναι υπεύθυνο για τις οικονομικές εξελίξεις. Από τη μια δηλαδή έχουμε περιβάλλον, από την άλλη έχουμε οικονομικές εξελίξεις. Είμαστε πεπισμένοι εμείς ότι αυτή η διάκριση ε, θα βοηθήσει να διασφαλιστεί η επιτυχία του συμβασμού στον οποίο έχουμε καταλήξει με την οδηγία αυτή. Ένα άλλο ζωτική σημασία στοιχείο είναι το θέμα της αδειοδότησης. Υπάρχει συμφωνία για τις προϋποθέσεις που πρέπει να καλύπτουν οι επιχειρήσεις οι οποίες ε, ζητούν αδειοδότηση για εξόριξη πετρελαίου κτλ. Λέμε δηλαδή ότι όσοι υποβάλλουν αίτηση για αδειοδότηση πρέπει πριν αρχίσουν οι δραστηριότητες να δώσουν αποδείξεις για την οικονομική τους ευρωστία προκειμένου να είναι βιώσιμο το σχέδιό τους. Είναι πολύ σημαντικό για μας αυτό. Επιτρέψτε μου επίσης αγαπητοί συνάδελφοι να αναφέρω ότι η πρόταση αυτή για οδηγία απευθύνεται σε όλες τις χώρες μέλη. Υπάρχουν ε, φυσικά πολλά επιχειρήματα ιδιαίτερα από χώρε όπω είναι Λουξεμβούργο, Αυστρία κτλ. που λένε με εμά δεν μα αφορούν, εμεί δεν έχουμε offshore δραστηριότητε, δεν έχουμε θάλασσα. Γνωρίζουμε όμω ότι υπάρχουν επιχειρήσει οι οποίε εδρεύουν, έχουν ε, τη διοικητική του έδρα σε τέτοιε χώρε, στην εδωχώρα δηλαδή. Οπότε για να υπάρχει ισορροπία και συμμεταχείριση, θεωρήσαμε ότι αυτή η οδηγία πρέπει να καλύπτει όλες τις χώρες. Οπότε και τέτοιες χώρες στην ενδοχώρα να πρέπει να ενσωματήσουν τουλάχιστον ε, τα ελάχιστα στοιχεία αυτής της οδηγίας στην εθνική τους νομοθεσία. Τέλος, κύριε Σαρτόρη, πρόκειται για την εγκληματική διάσταση. Ξέρουμε ότι είναι κάτι που έχει απασχολήσει πολλές φορές το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καταλήξαμε σε ένα συμβασμό, ε, συμφωνήσαμε τελικά με τον ορισμό που αποφάσισε στα τέλη του 2014 να ξαναδεί το Συμβούλιο, προκειμένου η οδηγία αυτή να εμπίπτει και στα πλαίσια της οδηγίας για την εγκληματική ευθύνη. Συμφωνήσαμε με την πρόταση αυτή. Του χρόνου θα δούμε τι συνέχεια θα δοθεί και τι άλλα στοιχεία θα έχει να μας δώσει η Επιτροπή για το θέμα της εγκληματικής ευθύνης. Τώρα το θέμα της ενσωμάτωσης και της εφαρμογής, όσον αφορά τις προθεσμίες δηλαδή, πρέπει να ξέρετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις έκανε λίγο πιο μικρές τις προθεσμίες αυτές, αλλά πιστεύουμε ότι είναι απόλυτα λογικό για τις επιχειρήσεις να μπορέσουν να προσαρμοστούν. Αυτά, κυρία Πρόεδρε, είναι τα κύρια στοιχεία του συμβιβασμού αυτού στον οποίο καταλήξαμε και πρέπει να ξέρετε ότι είμαστε πεπισμένοι πως οι περισσότεροι εδώ πέρα συμφωνούν με αυτή. Ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες αυτές που μας δώσατε. Τώρα, το σημείο 9, είπαμε ότι η συζήτηση με την κυρία Άννα Γένσεν, ειδική συγγήτρια, αναβάλλεται για τις 24 και 25 Απριλίου. Συνεπώς, διακόπτουμε. Αύριο το πρωί στις 9 θα αρχίσουμε πάλι και στις 5.30 θα αρχίσει η συνεδρίαση των συντονιστών. Χρειαζόμαστε χρόνο για να καταφέρουμε να τους φέρουμε και όλους εδώ. Λοιπόν, 5.30 οι συντονιστές. Οι υπόλοιποι αύριο το πρωί στις 9 εδώ.